Σας παρακαλώ καθίστε αρκετά σύντομα. Σύμφωνα. Βάση ε, της πράξης της 20 ης Φεβρουαρίου για την εκλογή των βουλευτών ε, με καθολική άμεση ψηφοφορία κηρύσω την έναρξη της πρώτης ε, Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις εκλογές.